για αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 70α του κανονισμού για την ε, έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και την εντολή για τρεις νομοθετικές διαβουλεύσεις. Η σειρά αυτών των οι, έχουν ε, μεταφραστεί στις γλώσσες και μπορούν να ε, αντληθούν από εσά από το διαδίκτυο. Θεωρείτε ότι εγκρίνονται εκτό αν μια κοινοβουλευτική ομάδα ή 40 μέλη μέσα σε προθεσμία 48 ωρών δεν θα θέσουν έτοιμα για συζήτηση και ψήφιση θα έχουμε τις νέες διαδικασίες για τις επιθυμίες για την πρώτη ανάγνωση, συμφωνίες για πρώτη ανάγνωση. Seance on direct. Μπορούν άμεσα να αντιληθούν από εκεί αυτά τα αιτήματα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Αν μέχρι 48 ώρες δεν θα υπάρξει από κάποια κοινοβουλευτική ομάδα ή από 40 μέλη έτοιμα για συζήτηση και ψήφιση, αυτό θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Αν όχι, αν δεν υπάρξει τέτοιο αίτημα, θα έχουν εγκριθεί αυτέ οι εντολέ. Την Τρίτη, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού, που τον πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψω 7 νομικέ πράξει ε, που υπόκεινται στην, έχουν εγκριθεί από την κανονική νομική, νομοθετική διαδικασία. Οι τίτλοι αυτών των νομοθετικών πράξεων θα εμφαίνονται στα πρακτικά τη σημερινή μα συνεδρίαση. Και περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη αυτή τη Συνόδου για την ημερήσια διάταξη